για την συστηματική μαζική δολοφονία των θρησκευτικών μειονοτήτων από τον IS, το Ισλαμικό κράτος. Η κυρία Μογκερίνη όμως δεν έχει έρθει ακόμα. Οπότε... Α, ωραία. Χαίρετε κυρία Μογκερίνη. If you want, you can start off. Παρακαλώ, ξεκινήστε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά χρειάστηκε να ασχοληθώ με κάτι το οποίο συζητήθηκε προγενέστερα. Θα ήθελα να σας πω καταρχήν ότι αυτή η συζήτηση σχετίζεται με ένα ζήτημα ύψης της σημασίας και σχετίστηκε με τη χτεσινοβραδινή συζήτηση, δηλαδή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την κατάσταση που αφορά τις αιρέσεις, γιατί ε, πολλές εθνότητες, μειονότητες και ιδιαίτερα θρησκευτικές μειονότητες συμβίωσαν στη Μέση Ανατολή. Και φυσικά ο σεκταρισμός υπάρχει ε, προαιώνια, αλλά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι τόσο ευάλωτη όσο σήμερα. Δυστυχώς όλοι προώθησαν το σεκταρισμό στα πλαίσια της κατάκτησης της εξουσίας και σήμερα βλέπουμε ότι δυστυχώς επικρατεί η μυσαλλοδοξία παντού. Και αυτό αφορά και τον ISIS και το Ισλαμικό κράτος, το οποίο χρησιμοποίησε τη μυσαλλοδοξία για να μπορέσει να προσελκύσει και να προσιλητήσει πολλούς. Πριν μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς να αντιμετωπίσουμε τις θρησκευτικές μειονότητες, θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Η βία δεν απειλεί μόνο τις μειονότητες και αυτό αφορά και την ΤΑΕΣ. Η ΤΑΕΣ σκότωσε πάνω από 100 ανθρώπους και απήγαγε επίσης εκατοντάδες την Νέη Σαλσόρ. Εάν δείτε τους αριθμούς, τον αριθμό των θυμάτων στις σειράξεις, βλέπουμε ότι η πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι. Αφορά την Συρία, το Ιράκ, όπως και την Ιγυρία και το Πακιστάν. Επίσης και στην Ευρώπη έχουμε θύματα ε, μουσουλμάνων. Και αυτό αφορά και τις τρομοκρατικές ενέργειες. Μιλάμε για ε, θύματα τα οποία θα πρέπει να υπερασπιστούμε. Αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα. Συμμετέχουμε όλοι και είμαστε ενωμένοι. Όμως, η κατάσταση των ε, ατόμων που ε, ε, βρίσκονται, που συμμετέχουν σε θρησκευτικές μειονότητες και ιδιαίτερα οι χριστιανικές κοινότητες, κουρδικές πόλεις, οι γυναίκες Γεζίτη, Σομπάτ, Δρούζη, Ασσύριοι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε καμία θρησκευτική μειονότητα. Μπροστά σε αυτή την ομότητα θα πρέπει όχι μόνο να καταδικάσουμε. Καταλαβαίνετε την απογοήτευσή μου κάθε φορά που θα πρέπει να προβώ σε μία δήλωση καταδίκης. Αυτό πρέπει να το κάνω γιατί δείχνει ότι δίνουμε σημασία σε αυτές τις μειονότητες και κοινότητες, αλλά η προφορική καταδίκη δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει έμπρακτα να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Πώς ε, υπερασπιστήκαμε τις μειονότητες στη Μέση Ανατολή. Καταρχήν, χρηματοδοτικό πακέτο προβάλλουμε συγκεκριμένη χρηματοδοτική υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη χρηματοδοτούν κατά πέντε δις την ε, Συρία. Είμαστε οι βασικοί δωρητές και είμαστε οι πρώτοι που υποστηρίξαμε τους Γεζίδη και τις χριστιανικές μειονότητες, τις επισκέφτηκα και τα Χριστούγεννα και αυτό αφορά και τους Κούρδους στο Κομπάνι. Τα χρήματα αυτά βοηθούν έτσι ώστε να ε, μπει στο κανάλι της ζωής αυτή η περιοχή που απελευθερώθηκε από το Νταές, από το Ισλαμικό κράτος. Μιλάμε ότι θα πρέπει οι να παραμείνουν στη γη τους, στη γη όπου ζουν εδώ και αιώνες. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για την Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορά την ανεξιθρησκεία και την πρόθεσή της και σημαίνει ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την κατάλληλη νομοθεσία και στη Συρία και στο Ιράκ όσο συνεχίζεται η συζήτηση είναι δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον σε μια μεταπολεμική κατάσταση. Το γνωρίζω πολύ καλά. Θα πρέπει όμως να έχουμε κατά νου ότι ο μακροχρόνιος στόχος είναι η ειρηνική δημοκρατία, χωρίς αποκλισμούς. Και αυτό θα πρέπει να γίνει ε, ειρηνικά, αν θέλουμε ένα καλύτερο αύριο. Θα ήθελα να είμαι ιδιαίτερα ειλικρινής. Οι πόροι είναι ανεπαρκής. Τα ανθρωπιστικά προγράμματα έχουν, δεν έχουν υποστηριχθεί όπως θα έπρεπε το 2015. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει το 2016 και εργαστήκαμε σε αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ανθρωπιστική βοήθεια και θα ήθελα να σας πω ότι βασιζόμαστε στο Κοινοβούλιο για να μας βοηθήσει και φέτος. Θα πρέπει να δεσμευτούμε απόλυλα στη σύσκεψη του Λονδίνου με συμμετοχή του Κουβέι, της Γερμανίας, της Βρετανίας και άλλων κρατών το Φεβρουάριο, έτσι ώστε να είμαστε οι βασικοί δωρητές. Επίσης, θα πρέπει να εγγυηθούμε την δικαιοσύνη, τη λογοδοσία. Αυτό είναι ένα βασικό βήμα προς την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή η οποία συλλέγει στοιχεία για ε, μελλοντικές ποινικέ διώξεις. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει πολιτική και οικονομική υποστήριξη και από την κοινωνία των πολιτών για τη λογοδοσία. Ζητήσαμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να προσάγει τη Συρία στο ε, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να θεωρηθούν αυτές οι πράξεις της ΝΤΑΕΣ γενοκτονία. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή των περιφερειακών φορέων και διεθνών οργανώσεων, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υποστήριξει τις μειονότητες στη Μέση Ανατολή. Από την απαρχή της κρίσης ήρθαμε σε επαφή με τους μουσουλμάνους εταίρους για την επίλυση του ζητήματος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνεισφέρουμε για την κατάλυση της ΔΑΕΣ, αλλά όχι με στρατιωτικά μέσα καταδικάσουμε τα εγκλήματα της ΝΤΑΕΣ, αλλά αυτό θα πρέπει να αφορά και τη μουσουλμανική κοινότητα και τις μουσουλμανικές αρχές που είναι ο καλύτερος εταίρος μας. Προωθούμε τη συνεργασία με τις μουσουλμανικές κοινότητες για να καταπολεμήσουμε την θρησκευτική μυσαλλοδοξία και τους τελευταίους μήνες αναβάθμισα τη συνεργασία με την οργάνωση αυτή. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, δράση της Επιτροπής Διάβιας και το Συμβούλιο Ασφαλείας το όπου ε, συγκεκριμένα κράτη είπαν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα άρνηση κυρίας που έχουν στην δίκη της γενοκτονίας αυτής. Χαίρομαι διότι στηρίζεται αυτή η στάση από όλα τα μέλη των Ηνωμένων Εθνών ή τα περισσότερα. Βρισκόμαστε στην εμπροστοφυλακή της διπλωματίας για να καταπολεμήσουμε την ΤΑΕΣ. Και θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζουμε και το έργο των Ιρακικών Αρχών και Συμφιλίωσης. Τέλος, στη Συρία βρισκόμαστε σε ένα στάδιο όπου τα εμπλεκόμενα μέρη θα προσπαθήσουν να βρουν το δρόμο τους για να ξεπεράσουν τον πόλεμο. Βεβαίως η πενταετής αιματοχυσία αποτελεί ένα επώδυνο παρελθόν, όμως δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να λάβουμε υπόψη την μεγάλη διαφοροποίηση της Μέσης Ανατολής θα πρέπει να υπάρχουν νέες δημοκρατίες χωρίς αποκλισμούς όπου όλοι να έχουν τα δικαιώματα που τους πρέπει. Παρά τις δυσχέρειες, οι μειονότητες στη Μέση Ανατολή δεν έχουν χάσει την ελπίδα τους. Ε, στο Αλέπο ένα μήνα πριν ε, άρχισε, άρχισαν οι πανηγυρισμοί ε, μέσα στα πλαίσια του ιοβιλέου της Καθολικής Εκκλησίας και άνοιξε η κεντρική πύλη της ε, τοπικής εκκλησίας. Πρόκειται για ένα δείγμα εμπιστοσύνης για ένα καλύτερο μέλλον. Σε μία πρόσφατη ε, συνέντευξη ο καθολικός επίσκοπος του Αλέπο είπε ότι ο Αλλάχ μπορεί να δώσει ζωή ακόμα και σε ένα μαύρο μυρμήγκι σε ένα ρογματόδι βράχο στην έρημο. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν δεν έχουν χάσει την ελπίδα. Εγώ δεν πιστεύω, όμως πιστεύω στο δικαίωμα όλων να ζουν σε κατάσταση ειρήνης. Πιστεύω στη διαφορετικότητα όπου να διαφυλάσσεται ταυτότητα των ανθρώπων, η ιστορία τους, το παρελθόν και το μέλλον τους, οι ελπίδες και οι φιλοδοξίες τους. Αυτή είναι η δύναμη της ανοιχτής κοινωνίας, η δυνατότητα συμβίωσης και αυτό είναι και η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής. Δεν μπορούμε να τους απογοητεύσουμε. Ο μόνος τρόπος για να μην γίνει αυτό θα είναι να επιζητήσουμε μια πολιτική λύση στην κρίση. Το συζητήσαμε αυτό χτες το βράδυ. Εδώ να μην υπάρχει μισαλοδοξία, να επιληθούν οι θρησκευτικές διαφορές και να υπάρξει εθνική συμφιλίωση. Οι φίλοι μας στη Μέση Ανατολή δεν έχουν χάσει ελπίδα. Εάν ε, τους λαμβάνουμε υπόψη, θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη. Και ας μην απογοητευτούμε ούτε εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Μογκερίνη. Περνάμε στη συζήτηση. Ε, ξέρετε ότι έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο και εδώ η βοηθός μου είπε ότι δεν θα υπάρχουν καθόλου μπλε κάρτες. Νομίζω ότι είναι σωστό. Λοιπόν, ο κύριος Αντάκτους για 1,5 λεπτό. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω την είπατε εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη για τη σημαντική δήλωσή της. Οι χριστιανοί στο Ιράκ και τη Συρία αντιμετωπίζουν καθημερινά καταστάσεις απαγωγών, βιασμών, βασανιστήριων και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους. Συνολικά ο αριθμός των χριστιανών έχει μειωθεί πάρα πολύ. Ο χριστιανισμός ε, και η τόπη λατρείας και όλα τα χαρακτηριστικά του εξαλείφονται. Άρα είναι απόλυτα αναγκαίο να σταματήσουμε το Ισλαμικό κράτος. Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα αναφέρεται ότι διαπράττονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δυστυχώ η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη. Το ISIS ε, είναι ένοχο για τα πιο αποτρόπαια, τα πιο άθλια εγκλήματα όπως τα ορίζει το Διεθνές Δίκαιο και πολλοί από τους ε, εξέχοντες δικηγόρους και νομομαθείς τονίζουν ότι αυτή η συνεχιζόμενη καταπίεση ε, ανταποκρίνεται ακόμη και στον πιο αυστηρό ορισμό της γενοκτονίας. Το Δεκέμβριο ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας είπε ότι οι διώξεις των χριστιανών έχουν υποτιμηθεί και δεν έχουν αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Μογκερίνη, αξιότιμοι συνάδελφοι, αυτό πρέπει να αλλάξει. Για να βοηθήσουμε τα θύματα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα αποκατάστασης και συμφιλίωσης έχουμε ιστορική ευθύνη να ευχαριστώ πολύ κύριε Αντάκτουσον, λέει ο πρόεδρος, 1,5 λεπτό τώρα, ο κύριος Βάιντενχολτσα. Εδώ πολύ συχνά έχουμε ασχοληθεί με τον ΝΤΑΕΣ, με αυτή την ε, νοοτροπία του θανάτου. Το ΝΤΑΕΣ καταστρέφει οτιδήποτε δεν είναι σύμφωνο με την απόλυτα άκαμπτη προσέγγιση της. Όλους τους πάντους, τους Αλεβίτες, τους Χριστιανούς, τους Σουνίτες, τους Σίτες, όλους αυτούς τους ε, διώκει. Δύο φορές εδώ σώμα έχουμε ασχοληθεί με το θέμα των ασυρίων χριστιανών και των γυναικών των Γεζίτη. Σήμερα μάθαμε ότι τον Νταέσ κατέστρεψε το μοναστήρι ε, του προφήτη Ηλία κοντά στη Μοσούλ που είναι ή ήταν 1400 ετών. Πρέπει να συνεχιστεί αυτός ο αγώνας με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ούτως ώστε στο μέλλον να υπάρξει δημοκρατία, ανεξιθρησκεία και ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτή την περιοχή. Πρέπει από τώρα να ξεκινήσουμε την εργασία για να προωθήσουμε τη συμφιλίωση, να δημιουργήσουμε τη βάση για το μέλλον της περιοχής. Αλλά πρώτα απ' όλα χρειάζονται όλοι όσοι ακόμη είναι όμοιροι των τρομοκρατών αυτών τη βοήθειά μας. Πολλές εκατοντάδες ε, γυναικών γεζιντή που υποφέρουν. Τις αντιμετωπίζουν ως ε, εμπορεύματα γιατί είναι απλώς πηγή εισοδήματος. Τις πουλούν και σε χώρες με τις οποίες έχουμε εμείς οικονομικές σχέσεις όπως η Σαουδική Αραβία για τους ε, Ασυρίους. Έχουμε ζητήσει 25 εκατομμύρια δολάρια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βάντιν Χόλτσο, ο Πρόεδρος. Και τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Τάνοκ. Απογοητεύομαι γιατί μιλάτε για συστηματική δολοφονία, για κάτι που είναι γενοκτονία. Πέρσι ήρθα σε επαφή με ιρακικές χριστιανικές μειονότητες και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ε, γεζίτη διώκονται έτσι ώστε να εκδιωχθούν όλοι και όλοι οι μουσουλμάνοι. Αυτοί που δεν είναι Σουνίτες βεβαίως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές γυναίκες γεζίτη στην ουσία κρατούνται, έχουν βιαστεί και πολλούνται ως σκλάβες και το Ηνωμένο, τα Ηνωμένα Έθνη, η Επιτροπή Ανθρωπιστικών Δικαιωμάτων είπε ότι πρόκειται πραγματικά για γενοκτονία. Δεν μπορούμε να δίνουμε αυτή τη σήμανση σε αυτά τα εγκλήματα και θα πρέπει να ε, διωχθούν ε, οι επικεφαλής του ISIS και να... Κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε Τάνοκ, κύριε συνάδελφε Τάνοκ, κύριε συνάδελφε Τάνοκ, κύριε Τάνοκ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με εσάς, αλλά οι συνάδελφοι, οι διερμηνείς σας παρακαλούν να μιλάτε πιο αργά προσπαθώ να μην σας ε, διακόψω. Αλλά εσεί δεν αντιδράτε και μιλάτε όλο και πιο γρήγορα. Δεν είναι το να διαβάζετε σε, τέσσερα, σε μία ομιλία τεσσάρων λεπτών σε ένα λεπτό. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί αλλιώ οι διερμηνείς, οι διερμηνείς δεν μπορούν να συνεχίσουν. Εάν συνεχίσετε να μιλάτε με αυτήν την ταχύτητα θα σας πάρω τον λόγο. Με συγχωρείτε, δεν αποφασίζετε εσεί πώ θα μιλήσω. Και θέλω να κάνω έκκληση στον πρόεδρο Σούλτ. Είναι δεύτερη φορά που με σταματάτε στη μέση τη ομιλία μου. Ενώ μιλάω για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν πολύ καλά τα αγγλικά. Με ευχαριστώ πολύ. Θα σα διακόπτω όλο και πιο συχνά αν θέλετε. Και δεν είναι αλήθεια ότι μπορείτε να μιλάτε όσο γρήγορα θέλετε. Στην αίθουσα αυτή υπάρχουν κανόνε όπου λέγεται σαφώ ότι εάν οι διερμηνείς δεν μπορούν πλέον να κάνουν διερμηνία τότε πρέπει να διακοπεί όλη η συνεδρίαση. Δεν μπορείτε λοιπόν να μιλάτε όσο γρήγορα θέλετε. Και τώρα επόμενος ο συνάδελφος Νάρτ. Για πόσο χρόνο, εάν πρόκειται να μιλήσετε με κανονικό ρυθμό, δεν σας δίνω το λόγο λοιπόν. Όχι, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Νάρτ. Για πόσο χρόνο παρακαλώ ο ε, κύριος Νάρτ. Α, ωραία, ευχαριστώ. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη Μέση Ανατολή χωρίς να κατανοήσουμε τις διάφορες κοινότητες. Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την ε, περιοχή αν δεν κατανοήσουμε τον Εβραϊσμό ο οποίος εξαφανίστηκε καθώς και τις διάφορες χριστιανικές ε, κοινότητες Χαλδαίων, Ασυρίων, Καθολικών και Μαρονιτών. Το πρόβλημα, κύριοι, δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει με το Ισλαμικό κράτος. Οι χριστιανοί του Ιράκ έφυγαν, άρχισαν να αποχωρούν μετά από την εισβολή της Αμερικής στο ε, Ισραήλ. Όλο ένα και αποχωρούν χριστιανοί. Η Βικλέμ που ήταν καταρχήν χριστιανική πόλη, τώρα έχει μία μικρή μειοψηφία χριστιανών, διότι η ζωή είναι αβίωτη και γιατί θα πρέπει να υπάρξει προστασία αυτών των μειονοτήτων σε κλειστούς χώρους. Το ίδιο έγινε και με τους Δρούζους και με τους Γεζίτη. Αυτό αφορά τους Αλαουίτες, τους Μαρονίτες, τους Σουνίτες και τους Σιήτες. Έχουμε να κάνουμε με θύλακους, με πλέον και αυτό αποτελεί τραγωδία. Γιατί αν δεν είμαστε αλληλέγγυοι, τουλάχιστον ας είμαστε αρκετά εγωιστές. Υπάρχει μια ισχυρή χριστιανική κοινότητα στη Μέση Ανατολή και αυτή, αυτό είναι το καλύτερο σημείο επαφής, η καλύτερη γέφυρα επαφής. Αυτό ίσχυε και με την Βοσνία, όπου όμως από όπου αποχώρησαν οι χριστιανοί. Δεν χρειάζεται να καταδικάζουμε με τα φυσικά. Δεν τους δώσαμε τίποτα, ούτε καν ελπίδα σε όλες αυτές τις χριστιανικές μειονότητες. Ευχαριστώ, συνάδελφε Νάρτ. Διαδικαστικό, παρακαλώ. Εάν ακούσετε την διερμηνία θα καταλάβετε ότι ήδη είπατε σας έδωσα ήδη το λόγο. Εάν ακούγατε τη διερμηνία θα το είχατε ακούσει. Έχετε το λόγο. Ναι, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Εντάξει, θα μιλήσω αρκετά αργά για να με καταλάβετε. Σας ευχαριστώ. Για δεύτερη φορά δείχνεται ασέβεια, έλλειψη σεβασμού απέναντι στον συνάδελφο. Τον διακόπτεται, ενώ μιλάει για πολύ σημαντικά θέματα. Πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη. Θα το πω στον πρόεδρο. Είναι μια ε, πολιτική η οποία δεν είναι σοβαρή απέναντι στον συνάδελφο. Ελπίζω να τα είπα αρκετά αργά για να με καταλάβατε. Και να με καταλάβατε δεν χρειάζεται να ενημερώσετε το Προεδρείο, θα τους το πω εγώ. Γιατί υπάρχει πολλή προϊστορία και προσπαθώ πάντα μέσω του μικρού μου σφυριού να κάνω στον κύριο Τάνοκ να καταλάβει ότι μιλάει πολύ γρήγορα. Εδώ έχω ένα κόκκινο φωτάκι. Δεν είμαι καθόλου υπεροπτικός. Και αν ε, συνεχίζει να μην αντιδρά ο κύριος Τάνοκ, τον διακόπτω. Και επειδή καθόλου δεν έκανε προσπάθεια να συμμορφωθεί, του πήρα το λόγο. Όλα αυτά είναι απόλυτα σύμφωνο με τον κανονισμό και θα ε, συμφωνήσει που πιστεύω το Προεδρείο. Για το θέμα αυτό, το διαδικαστικό, δεν θα το συζητήσω, θα το υποβάλω στο Προεδρείο. Επόμενος ο Σνάλφο Λου Αρίκ, για 1,5 λεπτό. Ο Ισλαμικό κράτος ε, και η συμμαχοί του απορρίπτουν τις ανθρώπινες αξίες, απορρίπτουν τη σκέψη ε, κρύβονται πίσω από το παραβάν μιας ε, θρησκείας την οποία βρωμίζουν σκοτώνοντας ε, τους πάντες, τους δημοκράτες, ό,τι δεν του μοιάζουν, τους μουσικούς, τους Κούρδους, τις ε, θρησκευτικές μειονότητες. Ε, σκοπίσουν παλού αίμα ε, στους ε, χριστιανούς, τους γεζίτες, τους αλαουίτες και τα βασικά θύματα αυτών των φασιστών είναι οι μουσουλμάνοι. Θα πρέπει να τους καταπολεμήσουμε αμήλικτα. Είναι τέρατα. Αυτό δεν πρέπει όμως να μας κάνει να μην σκεφτούμε τις πηγές και τις αιτίες που κατασκεύασαν αυτό, το, αυτή την τρομοκρατία. Ε, η κουλτούρα του νόμου του πιο δυνατού. Ε, το, το πετρέλαιο, οι πόλεμοι, οι θεσμοί θα πρέπει να δράσουν για να προστατεύσουν τις θρησκευτικέ μειονότητες, να μειωθεί ο, ο εγκληματικός μηδενισμός του Ισλαμικού κράτους και να βρεθεί ένα νέο πλαίσιο ευρωμεσογειακό εταιρική σχέσης για μία ε, ανάπτυξη ανθρώπινη όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία ε, Βαλέρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι επιθέσεις απέναντι στι σκεφτικές μειονότητες ε, παντού έχουν ε, αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Απέναντι στους Ασσύριους, ε, στους Χριστιανούς, σε οποιονδήποτε δεν πιστεύει στα ίδια με σένα, τον σκοτώνεις. Έχουν σκοτώσει χιλιάδες χριστιανούς και έχουν αναγκάσει πολύ περισσότερους να αφήσουν τις αιστείες τους. Έχουν καταστρέψει τόπους λατρείας των χριστιανών στο Ιράκ και σε άλλες χώρες επίσης. Υπάρχει εθνική κάθαρση, η ιστορία επαναλαμβάνεται, χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται, ο πληθυσμός των χριστιανών έχει μειωθεί στο ένα δέκατο αυτού που ήταν. Και μιλάμε για θρησκείες οι οποίες ήταν παρούσες για χιλιάδες χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να διερωτηθούμε τι, σημαίνει, τι συμβαίνει σήμερα. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη ε, γενοκτονία, για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ε, και στο παρελθόν οι θρησκευτικοί πόλεμοι κατέστρεψαν θρησκείες. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει περισσότερη προσπάθεια, ούτως ώστε οι εμπλεκόμενοι να σταματήσουν τις, ε, τη δράση τους. Είδαμε φρικτές εικόνες στα ΜΜΕ πρόσφατα. Πρέπει να σταματήσουν αυτές οι επιθέσεις σε εθνικές μειονότητες επίσης. Ο καθένας θα πρέπει να έχει δικαίωμα να ζήσει στην πατρίδα του και μάλιστα με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Πάκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να θίξω το τραγικό θέμα των διώξεων των χριστιανών στα, στους καταβλισμούς προσφύγων. Αφού αποφεύγουν τις εφρικαλότητες που περισσότερο βλέπουμε μόνο στις τηλεοράσεις μας, πολλοί χριστιανοί αντιμετωπίζουν στοχευμένη ε, καταπίεση λόγω της πίστης τους ακόμη και στους καταβλισμούς των ΗΠΑ παντού στην Μέση Ανατολή και είναι σκανδαλώδες ότι αυτό το παραδείσαμε και στη Γερμανία. Οι οικογένειες που επιστρέφουν στο Ιράκ αντί να συνεχίσουν να αντιμετωπίσουν τις διώξεις και την καταπίεση από ριζοσπαστικούς Ισλαμιστές φανατικούς Ισλαμιστές στην Ευρώπη. Και αυτό για τους χριστιανούς που είναι αρκετά τυχεροί ώστε να φτάσουν μέχρι την Ευρώπη. Η καταπίεση σε αυτού του καταβλισμού σημαίνει ότι πολλοί χριστιανοί φεύγουν από αυτού του καταβλισμού και μόνο σε αυτού του καταβλισμού μπορούν να κάνουν αίτηση για να αναγνωριστούν ω πρόσφυγε. Είναι τόσο κακή κατάσταση που μόνο πολύ λίγοι χριστιανοί υποβάλλουν αιτήσει οι οποίες, ε, τις οποίες μετά τις ε, χειρίζεται ο Οργανισμός των Αμών Εθνών. Είναι απαράδεκτο αυτό, ενώ υποτίθεται πως είναι σε ασφαλές μέρος. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να εφίστανται διώξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. ενάμιση λεπτό. Ο κύριος Μάια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σχεδόν κάθε μέρα μαθαίνουμε τις ε, φρικαλιότητες του Ντάες. Πόσες φορές είναι τώρα που τα έχουμε συζητήσει για αυτό το Ισλαμικό κράτος. Τι μπορώ να πω. Οι τρομοκράτες σίγουρα γελάνε όταν μας ακούνε. Συζητάμε χωρίς ε, να έχουμε συγκεκριμένη δυνατότητα να βοηθήσουμε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Πριν από μερικές μέρες ακούσαμε ότι 300 στον Ταΐρ Ελζόρ δολοφονήθηκαν. Αλλά δεν κάνουν μόνο αυτό. Συστηματική βιασμή, ε, υποδούλωση, όλα αυτά είναι τμήμα του καθεστώτος βίας. Και αυτό κυρίως θίγει αυτούς που είναι ε, πιστοί άλλων θρησκειών, οι οποίοι δεν έχουν καμία προστασία. Στη Μοσούλη, για παράδειγμα, ένα Μία πόλη που έχει μια χριστιανική παράδοση 1600 ετών από το 14 δεν υπάρχει κανένας χριστιανός. Και αυτό έγινε μέσω δολοφονιών και εκδίωξης. Ας μην έχουμε καμία αυταπάτη αγαπητοί συνάδελφοι. Το Ισλαμικό κράτος δεν θα σταματήσει έξω από την Ευρώπη. Ήδη το διαπιστώνουμε δεν έχει σταματήσει. Είδαμε τι έγινε πέρυσι. Και ο διακηρυγμένος στόχος τους είναι ακόμη και η Δύση να μην έχει χριστιανούς. Αυτές οι μαζικές δολοφονίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με απόλυτη αποφασιστικότητα. Λόγια δεν θα αρκέσουν. Ευχαριστώ, Σνάλφε Μάιερ. Ένα λεπτό. Η κυρία Ντότζ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα. Είναι σωστό εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο που έχουμε την ειρηνική ε, δημοκρατική εκπροσώπηση στα κράτη-μέλη να είμαστε ενωμένοι και να κατα δικάσουμε τις μασικές δολοφονίε θρησκευτικών μειονοτήτων από το Ισλαμικό κράτος. Βλέπουμε ε, εικόνες από μαζικές δολοφονίε, ε, μαζικούς βιασμού, αποκεφαλισμού, κεφαλισμούς, ε, βαρβαρότητες από φανατικού ζυχαντιστέ. Όμως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει κάτι παραπέρα, κάτι παραπάνω, να αναγνωρίζει αυτή την, και να μιλήσει για αυτή τη βαρβαρότητα και να πει τι είναι, γενοκτονία, ε, κατά των χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων. Σήμερα το απόγευμα ε, παρακολούθησα την παρουσίαση που έγινε ε, για εκείνες τις χώρες που αντιμετωπίζουν δίωξη χριστιανοί. Και βλέπω ότι οι διώξεις κάτω των χριστιανών αυξάνεται συν το χρόνο. Εκτιμάται ότι πριν από τον πόλεμο στη Συρία 400.000 ε, χριστιανοί ήταν στο Αλέπο. Σήμερα είναι 6.000 μόνο. Ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. 1,5 λεπτό η κυρία Αλιού Μαρή. Κυρία Υπατή εκπρόσωπε, στην σύμβαση της 9ης Δεκεμβρίου του 48 αναφέρει ως γενοκτονία όλες τις πράξεις που θέλουν να οδηγήσουν στον εκμηδενισμό κάθε ε, εθνικής, εθνοτικής ή θρησκευτικής ε, μειονότητας. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για χριστιανούς, αλλά εντάσσονται και οι χριστιανοί στα πλαίσια της γενοκτονίας. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τον ΙΕ να αναγνωριστεί αυτή η γενοκτονία. Γιατί δεν πρόκειται για μία λέξη. Έχει ένα συγκεκριμένο νομικό ε, σημασιολογικό περιεχόμενο και έχει βεβαίως και διπλωματικές προεκτάσεις. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία δεν πρόκειται ε, μόνο για μία, ε, έναν πόλεμο με βάση το δίκαιο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και όπλα, αλλά και το δίκαιο και η δικαιοσύνη για να υπερασπιστούμε τις μειονότητες, αλλά ιδιαίτερα τους χριστιανούς, γιατί έχουν μείνει μόνοι. Εμείς που μιλάμε για τις χριστιανικές ρίζες της Ευρώπης, φέρουμε μια συγκεκριμένη ευθύνη έναντι αυτών. Ευχαριστώ κυρία Λιωμαρία. μισή λεπτό. Ο συνάδελφος Καν. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την ύπατη εκπρόσωπο για τις δηλώσεις της επί του θέματος. Οι άνθρωποι στη, στο Ιράκ και στη Συρία βασανίζονται και φωνεύονται από το Ισλαμικό ε, κράτος. Γιατί όποιος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όποιος σκοτώνει κάποιον ε, είναι σαν να έχει σκοτώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και όποιος διασώζει κάποιον είναι σαν να έχει διασώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το Ισλαμικό κράτος έχει καταστρέψει και την πολιτιστική κληρονομιά μεταξύ άλλων, πέρα από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς το Ισλαμικό κράτος θέλει να εξοντώσει τις θρησκευτικέ μειονότητες που επέζησαν εδώ και αιώνες. Ενώ το Κοράνι λέει ότι δεν υπάρχει εξαναγκασμός στη θρησκεία, το Ισλάμ όπως το ορίζει το Ισλαμικό κράτος δεν απορρίπτει αυτή τη θεωρία. Εμείς θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις μειονότητες της Μέσης Ανατολής έτσι ώστε να δεχτούμε τη διαφορετικότητα. Ο καθένας διαθέτει θεμελιώδη δικαιώματα ανεξάρτητα από τις πεπιθήσεις και την εθνότητά του. Θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με τα θύματα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο συνάδελφος Λεγκούτκο. Ευχαριστώ. Οι συστηματικές μαζικές δολοφονίες δεν είναι επίσημη πολιτική ορολογία. Η σωστή λέξη είναι γενοκτονία. Στο νόμο δεν υπάρχει αυτή η έννοια συστηματικές μαζικές δολοφονίες, ενώ η γενοκτονία είναι συγκεκριμένη νομική έννοια. Έχει νομική έννοια. Σας παρακαλώ κυρία Μογκερίνη να χρησιμοποιήσετε αυτό τον όρο. Τον είπατε μια φορά να το λέτε συνέχεια ποιοι είναι θύματα τη γενοκτονία ναι, οι θρησκευτικέ μειονότητε και οι μουσουλμανικές, αλλά πρώτα απ' όλα οι χριστιανοί. Γιατί να το μην το πούμε και να το επαναλάβουμε συχνά. Και να το επαναλαμβάνετε, κυρία, είπατε εκπρόσωπε. πολλέ χιλιάδε χριστιανών δολοφονούνται κάθε χρόνο. Έχουν γίνει διάφορε γενοκτονίε στο παρελθόν και το απίθανο είναι ότι κάθε φορά που διαπράττονται δεν ε, αποκλήθηκαν γενοκτονία για λόγους πολιτικής ορθότητας. Αργότερα τις αποκάλεσαν έτσι, πολύ αργότερα. Ντροπή είναι αυτό. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε και αυτό, θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο κι εμείς. Ναι, υπάρχει γενοκτονία των χριστιανών σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Λεγκούτκο. μισή λεπτό. Ο κύριος Πέτεν. Η γενοκτονία των θρησκευτικών μειονοτήτων δημιουργεί δύο προβλήματα. Γιατί το κάνει το ISIS και τι μπορούμε να κάνουμε. Ο λόγο είναι ιδεολογικό. Ορισμένοι λένε ότι το ISIS εκπροσωπεί μια διαστροφή του Ισλάμ. Στην πραγματικότητα αποτελεί μια κυριολεκτική ερμηνεία του Κορανίου. Το Κοράνι λέει ότι πρέπει να κάνουμε πόλεμο στους απίστους, να τους σκοτώσουμε τους απίστους και να τους κάνουμε να τρομάξουν, να τους τρομοκρατήσουμε. Το Κοράνι είναι υπέρ των σταυρώσεων, των αποκεφαλισμών και της ε, υποδούλωσης, της σκλαβιάς. Ακόμη και ο συστηματικός βιασμός των μη μουσουλμάνων γυναικών ε, ε, μπορεί να δικαιολογηθεί από τη σούρα του Κορανίου που λέει ότι ό,τι πάρετε το δεξί σας χέρι μπορείτε να το έχετε ως ιδιοκτησία σας. Αυτό είναι ένας, ένα είδος της μουσουλμανικής ε, ε, θρησκείας με βάση το οποίο οι μουσουλμάνοι έφτασαν μέχρι τη Γαλλία τον 8ο αιώνα πριν τους ε, αποθήσουν. Πώς μπορούμε να νικήσουμε το ISIS. Πρέπει να υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ της Δύσης και αυτών των Ισλαμικών χωρών που δεν θέλουν να ζουν κάτω από το βαρβαρικό καθεστώς του ISIS. Το ISIS χρηματοδοτείται και φοδιάζεται από κάποιους πρέπει να σταματήσει αυτό. Ο πολιτισμένος κόσμος, κύριε πρόεδρε μου είπατε ότι έχω 1,5 λεπτό. Μου είπατε 1,5 λεπτό. Α, ευχαριστώ. Α, ωραία ο πολιτισμένο κόσμο πρέπει να καταλάβει ότι μια κυριολεκτική ερμηνεία του Ισλάμ δεν έχει θέση στι φιλελεύθερε δημοκρατικέ κοινωνίε. Πρέπει να σταματήσει η μαζική μετανάστευση από τι Ισλαμικές χώρε και να προσπαθήσουμε να εντάξουμε αυτού που έχουμε ήδη εδώ. Και γιατί οι επικεφαλεί των χριστιανικών εκκλησιών δεν αναγνωρίζουν ότι έχουν μια δυνατότητα να προσελκύσουν και να κάνουν μια ιδεολογική εκστρατεία για να προσελκύσουν του μουσουλμάνου Ευρώπη στο χριστιανισμό. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ενάμιση λεπτό ο κύριος Τζιμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τις διώξεις των χριστιανών εδώ. Σύμφωνα με το Open Doors, πάνω από 100 εκατομμύρια χριστιανοί διώκονται. 105.000 χριστιανοί πεθαίνουν κάθε χρόνο και η πιο διωκόμενη ομάδα είναι οι χριστιανοί. Υπάρχουν φυσικά και διώξεις άλλων ε, θρησκευτικών μειονοτήτων, αλλά η κατάσταση γενικά είναι φρικαλέα. Αυτά που κάνει το Ισλαμικό κράτος ε, στην ε, Αφρική, στη Μέση Ανατολή, δεν είναι απλώς διώξεις, είναι γενοκτονία. Οι χριστιανοί είναι θύματα, οι περιουσίες τους καταστρέφονται η χριστιανική κληρονομιά καταστρέφεται, είναι αναγκασμένοι να προσυλλητιστούν στο Ισλάμ, τους παίρνουν τα όργανα του σώματός τους και τα χρησιμοποιούν σε ένα λαθρεμπόριο οργάνων. Έχουμε λάβει πληροφορίες από μη κυβερνητικές οργανώσεις και από διάφορες θρησκευτικές και εκκλησιαστικές οργανώσεις για κάτι τέτοιο. Αυτό που με το όνομά του το πράγμα. Είναι γενοκτονία. Και άλλες θρησκευτικέ μειονότητες και μουσουλμανικές μάλιστα μειονότητες, οι γεζίντι και άλλες μειονότητες και αυτές είναι θύματα. Και αυτές ε, πάσχουν. Θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που κάναμε μέχρι τώρα. Είναι καθήκον μας, είναι το καθήκον του πολιτισμένου κόσμου αυτό. Ευχαριστώ κύριε Ενάμιση του Σάντρος Παντσέρη. Ευχαριστώ. Πολυάριθμες εκθέσεις δείχνουν ότι η βία κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Ιράκ και στην Συρία, Χριστιανοί, γεζίδι, Τουρκμένοι και άλλες μικρές κοινότητες έχουν μειωθεί δραματικά στις περιοχές που ελέγχει το ISIS. Τα εδάφη ε, στην πραγματικότητα ε, εξαφανίζει ε, άτομα τα οποία ανήκουν σε θρησκευτικέ μειονότητε. Ε, Είναι θύματα ε, δολοφονιών, ε, εμπορίου οργάνων κτλ. Και για να μην κάνουν να μην στο στον μουσουλμανισμό, στην πραγματικότητα φεύγουν από τις αιστείες τους. Ε, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, τον όρο γενοκτονία με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει να καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που, που διαπράττει το ISIS κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων ε, του Ιράκ και της Συρίας. Θα πρέπει η Κομισιόν επίσης να ε, προκαλέσει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για αυτό το πρόβλημα και να ασχοληθεί με την ανθρωπιστική κρίση θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα εάν δώσουμε ενιαία απάντηση στις συγκρούσεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή και αν υπάρχει πραγματική δέσμευση και των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών απέναντι στην επίλυση των προβλημάτων. Εν αναμονή κάνουμε ό,τι μπορούμε για να α, υπερασπιστούμε τις μειονότητες αυτές. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι χριστιανοί στη Συρία απειλούνται από το Ισλαμικό κράτος. Δυστυχώς η μειονότητα αυτή έχει συρρυκνωθεί σε αυτή την περιοχή. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποστηρίξουμε όλες αυτές τις ομάδες και με στρατιωτική εκπαίδευση. Τον Οκτώβριο του 2013 οι μαχητές οι μαχητές του στρατού της Συρίας προέβησαν σε μία αιματοχυσία δηλαδή όλοι οι μαχητές, ακόμα και οι υποστηρικτές ε, του ε, καθεστώτος, οδήγησαν σε αυτό το λουτρό αίματος. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει και εντός και εκτός των συνόρων μας. Δεν θα πρέπει να Ευχαριστώ, Σνάλφε Μπέλντερ. Ενάμιση λεπτό, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει λοιπόν εφόσον θέτουμε αυτά τα ερωτήματα να δίνουμε και απαντήσεις. Πρέπει να δούμε πώς έχει η πραγματικότητα. Πρόκειται ούτως ή άλλως για γενοκτονία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, να το αποδεχθούμε. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να δράσουμε, επειδή αντιμετωπίζουμε γενοκτονία. Με έχουν κουράσει όλες αυτές οι συζητήσεις για τις χριστιανικές μειονότητες για όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούω. Δηλώσεις, μόνο λόγια, μετά τίποτα. Καμία δράση. Το διαπίστωσα στο Ιράκ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανθρωπιστικά προγράμματα για να βοηθήσουν τους διοκόμενους. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε καλύτερα επιτόπου για να, για να υπάρξει περισσότερη βοήθεια επιτόπου από τοπικούς φορείς. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει όσους έχουν απομείνει από αυτές τις κοινότητες. Όσους έχουν απομείνει, γιατί παλιά ήταν ε, πολύ περισσότεροι, πάνω από ένα εκατομμύριο, όμως έχουν φύγει από την περιοχή. Πρέπει να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση, το λέμε συχνά αυτό. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν είναι εύκολο για αυτές τις θρησκευτικέ κοινότητες να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Όταν επισκέφθηκα την περιοχή, έμαθα ότι χρειάζεται συγκεκριμένη δράση επιτόπου εκεί για να μπορέσουν να αποφεληθούν από αυτή τη χρηματοδότηση. Εδώ θέλουμε να μα βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό. Η συνάδελφο Γκόμε. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους Κούρδους ε, Σουνίτες, Σιήτες, Αλαουίτες και όλες τις μειονότητες που υπέστησαν τη βία της Νταές. Αυτό το είδα στο ε, Ιράκ όπου νέοι γεζίδι έπρεπε να ε, απαλλαγούν από το ζυγό της ΔΑΕΣ. Υπάρχουν 4.000 σκλάβες, γυναίκες που έχουν πουληθεί ως σκλάβες αφού βιάστηκαν από τους ε, εκπροσώπους μαχητές του Ιρακικού κράτους. Αλλά όπως μας είπαν στο Ντοχούκ και στο Ερμπίλ, εάν θέλουμε να προωθήσουμε, να βοηθήσουμε τις θρησκευτικές μειονότητες, θα πρέπει να μπορούν να ζήσουν στη χώρα τους, στα σπίτια τους, όχι να καταφεύγουν στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή ανθρωπιστική βοήθεια και πρέπει να οργανωθούμε και να συντονιστούμε καλύτερα καταπολεμώντας την ΤΑΕΣ που είναι μια λερναία ύδρα. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωτίστως. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό, ο συνάδελφος Γιούρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η τραγωδία δεν θα είχε συμβεί εάν πριν από πολλά χρόνια θυμόμασταν ότι η ασφάλεια των χριστιανών στη Μέση Ανατολή θα έπρεπε να ήταν προτεραιότητά μας και να την προωθούμε στις πολιτικές μας. Όχι μόνη προτεραιότητά μας, αλλά μία από τις προτεραιότητές μας και ένα από τα πράγματα που συμπεριλαμβάνουμε σε όλες τις πολιτικές και στι διαπραγματεύσει με τους συμμάχους μας. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μία ανθρώπινη τραγωδία. Τώρα πρέπει να κινητοποιηθούμε, να κάνουμε κάθε προσπάθεια, αλλά να συνάγουμε και τα σωστά συμπεράσματα. Συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι εκεί λαμβάνει η χώρα μία γενοκτονία. Αλλά επίσης καταδικάζω και το μίσος κατά των χριστιανών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Σάνφε Γιούρεκ. Ενάμιση λεπτό. Ο Σάνφος Κέλλαν. Πέρσι περισσότεροι από 7.000 χριστιανοί δολοφονήθηκαν. Δύο χρόνια πριν ήταν 2.000. Οι χριστιανικές μειονότητες του Ιράκ έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες διώξεις ανά το κόσμο. Πέρσι είχαμε να κάνουμε με μία επέκταση αυτού του φαινομένου, μία τάση ε, όπου η μυσαλλοδοξία επικρατεί. Και θα πρέπει να δεχτούμε αυτή τη μορφή του ρατσισμού που δεν δέχεται τη συμβίωση όπου μιλάμε για όχι μόνο τρομοκρατικές πράξεις, αλλά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία. Τι πρέπει να γίνει. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρξει ανεξιθρησκεία, να οριστεί αυτό ως βασικός όρος σχέσεων με τρίτες χώρες. Επίσης να προσαχθούν οι υπέτειοι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη γενοκτονία αυτή. Επίσης η εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να αναμορφωθεί. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ανεξιθρησκεία που αποτελεί θέμενη αξία, διότι μόνο έτσι μπορούμε να εξουδετερώσουμε τον εξτρεμισμό. Επίσης, στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να υπάρχει ισότητα ως προς την, τις θρησκευτικές ε, πεπιθήσεις και αυτό που έχει σημασία είναι να επιστρέψουν όλοι στην πατρίδα τους. Ευχαριστώ ένα λεπτό. Η κυρία Κώστα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αλήθεια. Είμαστε μάρτυρες στις κατεχόμενες περιοχές από το Ισλαμικό ε, κράτος σε συστηματική δολοφονία και διώξεις. Αλλά απέναντι στους ε, χριστιανούς στην Ιγυρία, στη Συρία, στο Ιράκ έχουμε να κάνουμε με γενοκτομία με βάση τον ορισμό του ΟΗΕ. Γιατί οι χριστιανοί είναι η πιο διωκόμενη ομάδα. Ε, σχεδόν 100.000 ε, χριστιανοί δολοφονούνται ε, κάθε χρόνο και έχουμε και πολλούς οι οποίοι καταλείπουν τις αιστείες τους. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ε, συνέπεια στην, από την διεθνή κοινότητα. υπάρχει ε, τρομε, δίωξη από πλευράς του ΝΤΑΣ απέναντι σε αυτές τις κοινότητες. Είναι πραγματική πολιτιστική η κληρονομιά αυτή. Κυρία Μογκερίνη, εσείς είσαστε συνεπεί ε, στο επίπεδο της ανθρωπιστική βοήθειας, ε, σε επίπεδο διαλόγου που προωθείτε για την πρόληψη, για να ε, υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, να υπερασπιστούμε το δικαίωμα θρησκευτική. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία συνάδελφε. Ένα λεπτό, συνάδελφος Κρύπεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρία Υπατή εκπρόσωπη συνάδελφοι. Συζητάμε και πάλι τη συστηματική μαζική δολοφονία των, των θρησκευτικών μειονοτήτων από την Άση. Γιατί δεν τη λέμε. Γενοκτονία. Όπω είναι. Κάνω την ίδια ερώτηση με προηγούμενου. Οι χριστιανοί στη Συρία δολοφονούνται ή εγκαταλείπουν τι αιστείε του. Μόνο η μισή από το 1,25 έχουν μείνει και σε άλλε περιοχέ, το 80% περίπου έχουν εκριζωθεί. Αν δεν κάνουμε κάτι η κατάσταση ε, θα είναι ότι δεν θα μείνει κανεί. Και το ίδιο είναι με του Γεζίδι. Πολλέ εκκλησίε ε, καταστρέφονται ή γίνονται τζαμιά. Αυτό συμβαίνει στη Συρία και στο Ιράκ, αλλά και στην Τουρκία. Σα καλώ, κυρία είπατε εκπρόσωπε, να μα παρουσιάσετε συγκεκριμένα βήματα από την Κομισιόν για να το κάνετε αυτό περαιτέρω. Η απειλή αυτή είναι και εδώ στην Ένωση. Είδαμε του χριστιανού, του ε, καταβλισμού προσφύγων στην Ευρώπη να εφίστανται επιθέσει από άλλου πρόσφυγε λόγω τη πίστη του. Τι θα κάνει η Κομισιόν. Αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτή τη συστηματική μαζική δολοφονία και να δώσουμε σε αυτέ τι σχετικέ ομάδε ελπίδα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για γενοκτονία και να βοηθήσουμε τη δημοκρατική αυτοδιοίκηση στην βορειοανατολική Συρία, στην Ροτζάβα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σάλφε Κρίπεκ. 1,5 λεπτό ο Σάλφο Τατζάνη. Το 2020 στο Ιράκ και τη Συρία δεν θα υπάρχουν πλέον χριστιανοί, ούτε γεζίδι. Αυτό μας λένε οι προβολές. Είχε δίκιο η Χίλαρη Κλίντον όταν μίλησε για γενοκτονία, η πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε τη στάση αυτή της Χίλαρη Κλίντον, που θα είναι μάλλον και μελλοντική πρόεδρος τον είπα. Θα πρέπει να εισακουστούν αυτές οι προσπάθειες. Είναι ευπρόσδεκτες όλες οι πρωτοβουλίες, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να εισακουστεί ακόμα περισσότερα, διότι στη βία θα πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά. Η Ευρώπη υπάρχει γιατί πιστεύει στον άνθρωπο. Είναι μία ανθρωποκεντρική δύναμη. Αυτό μας επιβάλλουν και οι συνθήκες πέρα από τις αξίες μας. Μιλάμε για ανεξιθρησκεία. Υπάρχει συνεχής γενοκτονία των χριστιανών και των γεζίτη. Και η αντιμετώπιση αυτής της γενοκτονίας είναι προτεραιότητα, διότι διακυβεύονται οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικά θα έχουμε να κάνουμε με μια αδύναμη Ευρώπη που θα ασχολείται με τράπεζες και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ στον Αφιταγιάννη. Ένα λεπτό, η συνάδελφος Γκίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Υπατήκ Πρόσωπα. Η ΝΤΑΕΣ ε, συλλαμβάνει, φυλακίζει, βασανίζει και δολοφονεί ε, χριστιανούς και γεζίτη. Μόνο αυτή τη βδομάδα 400 απήχθησαν ή σκοτώθηκαν στη Συρία. Και το παλαιότερο χριστιανικό μοναστήρι στο Ιράκ ε, στην ουσία δεν υπάρχει πια. Εξαρθρώθηκε. Έχουμε να κάνουμε και με την ε, αλληλεπίδραση των Ταλιμπάν στην ΤΑΕΣ και θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει με τις ε, μειονότητες ο Ροπ Φλελόου από τα Midlands πίεσε ώστε οι ομότητες αυτές κατά των θρησκευτικών ε, μειονοτήτων γενοκτονία. Σας προτρέπω, σας προτρέπω και εσάς ως ύπατη να αντιμετωπίσετε το ζήτημα κατά αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί, να υπάρξει δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Πιετρόφσκι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Οι χριστιανοί είναι και η περισσότερο διοκόμενη μειονότητα. Το περσινό μας ψήφισμα τόνισε το γεγονός ότι 150.000 χριστιανοί αποτελούν αντικείμενο βίας και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις δολοφονίες του Ισλαμικού κράτους που καταστρέφει και τις εκκλησίες των χριστιανών που τους βασανίζει, τους ε, πνίγει, τους δολοφονεί οι πράξεις του Ισλαμικού κράτους αποτελούν γενοκτονία. Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει από πέρσι, όπως ζήτησε το Κογκρέσο, τον ΙΠΑ. Και βλέπουμε ότι και, το Ευρωπαϊκό, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ θα ήθελαν να μιλάμε για γενοκτονία πλέον. Και νομίζω ότι έτσι θα πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτές τις ομότητες. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό. Ο συνάδελφος Μιγιάν Μόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2015 ήδη εκφραστήκαμε επανειλημμένα για τις αποτρόπες επιθέσεις κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων στην ε, Μέση Ανατολή και την Αφρική. Στην ε, απόφασή μας του περασμένου Απριλίου είπαμε ότι οι χριστιανοί είναι η θρησκευτική κοινότητα που υφίσταται τι περισσότερες στον κόσμο και αυτό το είπαμε και σε άλλες εκδηλώσεις που κάναμε τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο. Όλοι οι θεσμοί πρέπει να ασχοληθούν ιδιαίτερα με την δραματική κατάσταση των χριστιανών, να τους βοηθήσουμε. Όπως υπόθηκε, είναι πολύ σημαντική η που συμπεριφορά του Ντάες και άλλων τοποκρατικών ομάδων έναντι των χριστιανών και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων. Έχουμε τις δηλώσεις του Αρχιπισκόπου του Μοσούλ, του Κύρκου και της Βαγδάτης για την καταστροφή των ε, τόπων λατρείας. Σήμερα, όπως υπόθηκε, είδαμε ότι καταστράφηκε κοντά στην Μοσούλη το μοναστήριο του Προφήτη Λία. Νομίζω ότι μειώνονται πάρα πολλοί χριστιανοί στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή είναι το 4% του πληθυσμού τη Μέση Ανατολή, ενώ πριν από ένα αιώνα ήταν γύρω στο 20%. Βεβαίω, η ήττα του Ντάε και η επίλυση τη ε, σύγκρουση στη Συρία θα βοηθούσε πάρα πολύ. 1,5 λεπτό είπατε, Πρόεδρε. Του τελευταίου μήνε ε, επανειλημμένα, η κυρία Μογκερίνη από πολύ διακεκριμένα βήματα είπε ότι θα έπρεπε να χαρακτηριστούν ως γενοκτονία αυτές οι ενέργειες. Θα ήθελα να μάθω την άποψή τη και την άποψη του Συμβουλίου. Δεν είμαι σίγουρο όμω ότι εκφράστηκε κατηγορηματικά. Γι' αυτό θέλω να δω ποια είναι η άποψή τη. Πρέπει οπωσδήποτε να μην υπάρξει ασυδοσία για τον ΤΑΕΣ. Τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει να εμπλακούν πολύ ενεργά στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Σάρφη Μιγιανμόν. Ενάμιση λεπτό η συνάδελφο Γκιαρντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι σήμερα υπάρχει αυτό ο Ισλαμικό ε, σε πολλούς τόπους για τους χριστιανούς η επιλογή είναι ή να προσελκυστούν ή να πεθάνουν ή να το σκάσουν. Μόνο στη Συρία 700.000 χριστιανοί εγκατέλειψαν τη χώρα τους. Αυτό σημαίνει ότι το 56% των χριστιανών φύγαν από τη Συρία. Ακόμα και στο Ιράκ είναι, έχουν αποδεκατιστεί. Είναι ελάχιστα τα στοιχεία, αλλά όλα τα στοιχεία ε, μονοσήμαντα μας λένε ότι οι χριστιανοί είναι η κοινότητα η πιο διοκόμενη στον κόσμο. Σε ορισμένε περιοχές όπως αναφέρθηκε, ούτε και η βοήθεια του ΟΗΕ δεν φτάνει στους χριστιανούς. Γιατί ε, τα στρατόπεδα των προσφύγων όπου βοηθάει ο ΟΗΕ ε, τα αποφεύγουν οι χριστιανοί γιατί φοβούνται να πάνε πραγματικά σε αυτά τα στρατόπεδα τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΗΕ. Ε, αισθανθήκαμε ε, ε, συγκίνηση όταν είδαμε τους αποκεφαλισμούς των κοπτών από το ISIS. Αλλά νομίζω ότι υποτιμούμε αυτή τη γενοκτονία. Θα πρέπει... Πώς θέλετε να την ονομάσουμε αυτή τη δίωξη μια τέτοια διάστασης όπου στη Βοσνία το, από το 1991 ε, μέχρι, μέσα σε 10 ε, χρόνια ε, ο αριθμός των χριστιανών μειώθηκε κατά 92%. Είναι γενοκτονία. Δεν είναι γλωσσικό το θέμα. Υπάρχει ένα φαινόμενο ε, που εντάσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ε, νομικό πλαίσιο και που ε, απαιτεί μία στρατηγική από τη διεθνή κοινότητα πολύ πιο έντονη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό τώρα ο συνάδελφος Βέντα. Ευχαριστώ. Διάφοροι συνάδελφοι ανέφεραν ότι οι τζιχαντιστές κατέστρεψαν και ακόμα ένα ιστορικό μνημείο, το μοναστήρι του προφήτη Λία στη Μοσούλη το λεγόμενο Ισλαμικό ε, είναι υπεύθυνο για την καταστροφή εκατοντάδων μνημείων. Οτιδήποτε ε, είναι κατά της δικής του ερμηνεία του Ισλάμ. Ε, διάφορες ε, ε, ξαφανίζονται. Οι χριστιανοί βασανίζονται, δολοφονούνται. Τα αγαθά τους τα παίρνουν. ο αριθμός των χριστιανών μειώνεται δραματικά. 2,5 εκατομμύρια ήταν παλιά και τώρα έχουμε 800.000 χριστιανού. Μέσα σε λίγα χρόνια μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου χριστιανοί. Η βία επίση πλήττει και του ε, Τουρκμένου, του Κούρδους, του Γεζίντι. Θα πρέπει να κάνουμε αποφασιστικά βήματα ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα ελεύθερη λατρείας και να καταδικάσουμε τις πράξεις του ISIS που θα πρέπει να τις ονομάσουμε ε, γενοκτονία και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ευχαριστώ, συνάδελφε Βέντα. Ένα λεπτό. Ο συνάδελφο Δίας Δεμέρα Γαρθία Κοσουέβρο. Θα πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη στα θύματα διωγμού. Και όπως ξέρετε την Τρίτη τα Ηνωμένα Έθνη μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Ανθρωπιστικής Δραστηριότητας μίλησε για γενοκτονία και αυτό αφορά και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Γι' αυτό, κυρία Μογκερίνη, συμμερίζομαι τις τέσσερις δράσεις που προαναφέρετε χρήματα, δικαιοσύνη, ε, διεθνής δέσμευση και διπλωματία. Χρειάζεται λοιπόν να απονεμηθεί, να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί όταν σταματήσει η τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ατιμορρησία. Και οι τρομοκράτες θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, ότι θα διωχθούν δηλαδή από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ότι θα δικαστούν και θα καταδικαστούν για τα εγκλήματά τους. Αυτό είναι και το καθήκον σας, να προωθήσετε αυτή τη δράση στο Διεθνές Ποινικό.

ότι οι χριστιανικές ε, μειονότητες έχουν μειωθεί κατά δύο τρίτα στη Συρία από το 2011 και μετά. Αυτό οφείλεται στην ολιγορία μας, διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπόρεσε να συμφωνήσει για να υπάρξει μία επέμβαση στη χώρα. Έτσι θα είχαμε αποφύγει και αυτή την ογκώδη και ολοένα και διονγκούμενη ροή στα σύνορα της Ευρώπης. Είτε μιλάμε για εγκλήματα είτε για γενοκτονία, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, δημιουργώντας μία ειδική διάρθρωση ασφάλειας και ανταλλαγής πληροφοριών. Να σταματήσουμε τη βαρβαρότητα. Ευχαριστώ. Η συνάδελφο Μανέσκου ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, τη συνάδελφο Αντάκτουσον και την ε, τη εκπρόσωπο την κυρία ε, Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε πλέον την δίωξη των Γεζίντι από την ΤΑΕΣ. Η σκλαβιά των Γεζίντι και οι βασανισμοί καθώς και οι βιασμοί θα πρέπει να θεωρηθούν γενοκτονία. Μετά τις δηλώσεις του Αλμπαγντάντι που είπε ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με τους ε, Γεζίδι ή τους Εβραίους και μετά το δόγμα προσιλητιστείτε ή ε, πεθάνετε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την φάση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα δύο τρίτα των χριστιανών έχουν αποχωρήσει από τη Συρία τα τελευταία πέντε χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν η διεθνής κοινότητα να δράσει άμεσα. Μετά το, τη Σρεμπρένιτσα και τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα θα πρέπει να πούμε never again. Ευχαριστώ ένα λεπτό η συνάδελφο Χιμένεθ Μπεθερίλα. Ε, νομίζω ότι μιλάμε για ελευθερίες, βαρεθήκαμε πια, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για ανεξιθρησκεία. Να μπορεί κανείς να δημιουργεί, να κάνει το σταυρό του και να μην πεθαίνει γι' αυτό. Δεν μιλώ μόνο για χριστιανοί, γιατί είμαι πολύ υπερήφανη που είμαι χριστιανή, αλλά υπερασπίζομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν μπορούμε να δεχτούμε τη συστηματική δολοφονία των χριστιανών από το Ισλαμικό κράτος. Βλέπουμε πια, ε, βλέπετε αυτές τις ε, φωτογραφίες ε, γυναικών γεζίδι που πολλούνται για 50 και για 100 ευρώ. Τα μικρά κορίτσια προς 100 ευρώ. Δηλαδή γίνεται λόγος για το γνωμικό προσιλητιστείτε ή πεθάνετε. Δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο. Τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν αυτή τη γενοκτονία. Τα θύματα μας κοιτάν στα μάτια. Κάτι πρέπει να κάνουμε και να το κάνουμε άμεσα. Ευχαριστώ. Ενάμιση λεπτό η κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε δολοφονίες, ε, διώξεις, το κάψιμο των εκκλησιών και των χριστιανικών συμβόλων. Ε, όλα αυτά σημαίνουν ότι οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή έχουν μία μόνο δυνατότητα. Ή θα πρέπει να μείνουν χριστιανοί, να παραμείνουν χριστιανοί, δύο δυνατότητες λοιπόν, ή να παραμείνουν χριστιανοί και να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους ή να αλλάξουν, να αλλαξοπιστήσουν για να επιζήσουν. Αυτό είναι το τρομερό έγκλημα. Είναι λοιπόν νομοτελειακό να, εξαφανιστούν πλήρως οι χριστιανοί του Ανατολή πριν εμείς πούμε ότι είναι γενοκτονία του Άσης αυτό πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι χριστιανοί ήταν 20% του πληθυσμού της Μέσης Ανατολής. Τώρα είναι μόνο 4%. Τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των χριστιανών στο Ιράκ πήγε από 1,4 εκατομμύρια σε 300.000 στη Συρία ο αριθμός μειώθηκε από 1,25 εκατομμύρια σε 500.000. Υπήρχαν 45 εκκλησίες στη Μοσούλη. Δεν υπάρχει καμία τώρα. Υπήρχαν 140 εκκλησίες ε, που καταστράφηκαν στη Συρία. Το παλιότερο μοναστήρι του Ιράκ που ήταν 1400 ετών και τώρα έχει ισοπεδωθεί. Δολοφονούνται, διώκονται χριστιανοί για να εξαλειφθούν. Πώς μπορούμε να ε, ερμηνεύσουμε αυτά που λέει το Άισι ότι θα κατακτήσουμε τις ε, περιοχές σα, θα πουλήσουμε τα παιδιά σας σκλάβους Αν δεν το επιτύχουμε εμείς, θα το επιτύχουν τα παιδιά μας. Οι χριστιανοί είναι η πιο διοκόμενη θρησκευτική κοινότητα παντού. Είναι θύματα γενοκτονίας. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση δείχνει ότι είναι ένα θέμα που αξίζει της πλήρους προσοχής μας. Στην ομιλία μου θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι οι θρησκευτικές μειονότητες συχνά δεν έχουν καμία ευκαιρία να ζήσουν μια κανονική ζωή. Μερικές φορές δεν μπορούν να ζήσουν καθόλου σε ορισμένα μέρη. Στην Κίνα, Φερρυπίν, οι χριστιανοί υφίστανται διακρίσεις επίσης. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι Φερρυπίν οι Εβραίοι στην Ευρώπη αισθάνονται πολύ άβολα Υπάρχουν πληροφορίε ότι οι Εβραίοι εγκαταλείπουν την Ευρώπη αυτή, σε αυτή τη φάση. Το οποίο δεν είναι καλό για την εικόνα μας. Αλλά η παρέμβαση για τις ζωέ των σκεφτικών μειονοτήτων ε, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, ιδίω στα εδάφη που είναι υπό την κυριαρχία του Ντάες. Είμαι πεπισμένο ότι η βία απέναντι στα θύματα λόγω της θρησκευτική πίστης είναι κάτι το οποίο απορρίπτουμε όλοι. Ε, το έχει δείξει η συζήτηση αυτή. Θα ήθελα επίση να τονίσω ότι το μοντέλο του δικού μας πολιτισμού που είναι ανοχή, μη διακρίσεις, τη δυνατότητα ειρηνική συνύπαρξης των διαφόρων θρησκειών και πολιτισμών στο όνομα αυτών των αρχών και για να υπάρξει δικαιοσύνη θα πρέπει να καταδικάσουμε την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Όχι απλά την καταδικάσουμε όμως. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη συνέχιση των δράσεων της διεθνούς κοινότητας. Και αν το να ονομάσουμε αυτές τις φρικαλαιότητες ε, γενοκτονία μπορεί να βοηθήσει αυτό, φυσικά το υποστηρίζω. Ευχαριστώ. Περνάμε στο ΚΑΤΣΤΙΑΕ τώρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώ έχουμε μεγάλη καθυστέρηση και έχω το διπλό αριθμό που έχω ζητήσει το λόγο από αυτό που θα μπορούσα να δώσω. Οπότε πρέπει να τονίσω ότι θα είναι μόνο ένα συνάδελφο από, από κάθε πολιτική ομάδα. Και από ό,τι ξέρω θα προσπαθήσουν να πάρουν το λόγο αυτοί που δεν έχουν πάρει συχνά το λόγο. Οπότε πρώτα απ' όλα δίνω το λόγο στην συνάδελφο Ζαμπόρσκα. Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπο. Η δράση της ΔΕΣ είναι κάτι το απαράδεκτο. Ε, θα πρέπει να αποκαλεστεί γενοκτονία. Θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει ένα ψήφισμα καταδικάζοντας τα βία εγκλήματα του Ισλαμικού κράτους και φυσικά ε, προσάγοντας τους υπευθύνους το διεθνές ποινικό δικαστήριο. Η κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ είναι παρόμοια με αυτή των σφαγών της Ρεμπρένιτσα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Εάν μιλάμε για γενοκτονία, τότε θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους χριστιανούς της Συρίας και του Ιράκ κατά των Σαλαφιστών. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Τώρα για ένα λεπτό ο συνάδελφος Τσαμπάσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το Ισλαμικό κράτος διαπράττει σφαγές στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία. Χιλιάδες χριστιανοί, Κούρδοι, Σιήτες είναι νεκροί. Το ξέρουμε όλοι μας. Και το συζητήσαμε πολλές φορές. Ε, εδώ και ένα χρόνο τα συζητάμε αυτά. Τι κάναμε όμως, τι πετύχαμε, τίποτα. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω το εξής. Το Ισλαμικό κράτος δεν κάνει πόλεμο με δηλώσεις. Με μεγάλα λόγια. Εάν δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο Ισλάμ, ε, είναι σαν να μην θέλουμε να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Η Τουρκία βοηθάει το Ισλαμικό κράτος, δίνει στη Συρία φάρμακα και όπλα. Θα πρέπει να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη γιατί αλλιώς θα κάνουμε τίποτα. Κυρία Μογκερίνη, θα πρέπει να υπάρξει ένα συμβιβασμό σε διεθνέ επίπεδο για στρατιωτικέ επιχειρήσει. Ευχαριστώ Λοιπόν, ο συνάδελφο ηλικιώτη τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε κυρία Μορκερίνη. Η τραγική κατάσταση με τι συνεχείς δολοφονίες και τι μαζικέ εξοντώσεις μελών θρησκευτικών μειονοτήτων από τον ISIS προσλαμβάνει ανεξέλεκτε διαστάσει. Χριστιανοί, οι Γεζίτοι, οι Δρούσοι, οι Ασσύριοι, όπω και τα μέλη άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων απειλούνται καθημερινά. Το ISIS έχει στόχο να του εξαφανίσει. Μιλούμε για γενοκτονία. Γι' αυτό δεν αρκούν τα ευχολόγια πρέπει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και να πάρουμε αποφασιστικά μέτρα. η ευρωπαϊκή ένωση δεν είναι άμυρη ευθυνών για τα όσα συμβαίνουν. με την ανοχή της ευρωπαϊκής ένωσης τόσο η γαλλία όσο και η γερμανία εξόπλιζαν τους τζιχαντιστές ενώ μέχρι σήμερα η ένωση γίνεται ουραγός των ηπα και των σχεδίων της για επαναχάραξη των συνόρων της ευρύτερης μέσης ανατολής συμβάλλοντας έτσι στην αποσταθεροποίηση της περιοχής. φτάνει η υποκρισία είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αιτίες που δημιούργησαν και ενίσχυσαν τον άισις να τερματιστούν οι ξένες επιβάσεις και οι πόλεμοι στον αραβικό κόσμο να στηρίξουμε έμπρακτα πρωτοβουλίες για ειρήνευση στη μέση ανατολή. Ευχαριστώ κύριε Σιλικιώτη. Και ο συνάδελφος Έκαρος τελευταίος διαδικασίας Catch the Eye. Θα ήταν σκόπιμο να ε, ρίψουμε το Ισλαμικό κράτος στη λίθνη εποχή. Δυστυχώς όμως έχουμε να κάνουμε με κυβερνήσεις των τόρις που στην ουσία υπερασπίζονται με νύχια και με δόντια μία πολιτική η οποία θα διαπραγματευτεί με αυτά τα ζώα του Άισις. Αυτό κάνουν οι εργατικοί. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτούς τους σατανιστές που ε, διακυβεύουν το μέλλον και την ελευθερία μας. Ευχαριστώ, συνάδελφε Έκα. Διαδικαστικό, ο κύριος Μάια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω ένα θεμελιώδες ερώτημα ε, για το πώς θα εφαρμόζεται τον κανονισμό. Άκουσα ότι κάθε ομάδα θα ληφθεί υπόψη. Το άκουσα. Δεν βλέπω όμως κανέναν κανένα να πήρε το λόγο από την ομάδα μου. Είπατε ότι πήρε το λόγο ένας μη εγγεγραμμένος. Είπατε ότι θα πάρει το λόγο κάποιος από τους μη εγγεγραμμένους. Πώς λοιπόν ε, εφαρμόζεται ο κανονισμό ε, συνήθως, τον εφαρμόζεται πολύ σωστά. Γι' αυτό σας παρακαλώ να πάρει κάποιος το λόγο και από τη δική μας πολιτική ομάδα. Γιατί αλλιώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ανακοινώσατε. Ευχαριστώ κύριε Μπαμάιρα. Νομίζω ότι και αυτή τη φορά σωστά ερμήνευσα τον κανονισμό. Ε, όταν είπατε ότι δηλώσατε ε, την παρουσία σας νόμιζα ότι θέλατε μπλε κάρτα και είχα πει δεν θα πάρουν καθόλου μπλε κάρτες. Δεν ακούμε τι λέει ο κύριος Ομπερμάιερ. Κύριε Ομπερμάιερ, σας δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ. Είστε πολύ γενναιόδωρος πρόεδρε. Θέλω να συμφωνήσω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε σήμερα αυτές τις μαζικές δολοφονίες, τα εγκλήματα του Άσης, ε, πραγματικά να το συζητήσουμε. Γιατί δεν αρκεί μόνο να το συζητήσουμε ωστόσο. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιθέσεις κατά αυτών των θρησκευτικών κοινοτήτων συμβαίνουν και στα δικά μας κέντρα υποδοχής προσφύγων. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη και αποφασιστική δράση από τις χώρες όπου υπάρχουν καταβλισμοί προσφύγων. Υπόθηκε ήδη ότι είναι γενοκτονία αυτό. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να τιμωρήσει τις χώρες που είναι υπεύθυνε για αυτά. Για παράδειγμα, τη Ειδική Αραβία, τα Εμμυράτα, που εδώ και πολύ καιρό δεν κάνουν τίποτα. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει να εξαπατάται. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε στο πλευρό των καταπιεσμένων και ιδιαίτερα στο πλάι των χριστιανών αδερφών μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ομπεμάιλε και ο Πρόεδρος. Έληξε η διαδικασία KFCI και στο τέλος της συζήτησης θα μιλήσει από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Επίτροπος κυρία Μογκερίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με το θέμα του ορισμού της γενοκτονίας. Δεν απέφυγα να το αναφέρω αυτό το θέμα στην αρχική μου παρέμβαση γιατί είμαι απρόθυμη, αλλά γιατί ο ορισμός ε, της γενοκτονίας ε, πρέπει να πληρεί συγκεκριμένα νομικά κριτήρια. Και αυτή η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί στα αρμόδια θεσμικά όργανα που είναι ο ΙΕ. Αυτό είναι το σωστό πλαίσιο. Η μόνη αναφορά μέχρι στιγμής στη γενοκτονία σε έγγραφα του ΟΗΕ είναι αυτό που έγινε πέρυσι στις 13 Μαρτίου του 2015 στην έκθεση του γραφείου του ΙΠΑ του εκπρόσωπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα για, τα, για την κατάσταση στο Ιράκ και για τις παραβιάσεις του Ισλαμικού κράτους ε, στο Ιράκ ε, και στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για βίες πράξεις κατά πολιτών λόγω του ότι ε, ανήκουν σε μια εθνική ή θρησκευτική ομάδα. Αυτή η έκθεση λέει ότι κάποιες από αυτές τις ε, πράξεις, ε, τις βίες πράξεις, μπορεί να αποτελούν γενοκτονία στην περίπτωση των Γεζίτη και, άλλον, και άλλη βία μπορεί να αφορά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή εγκλήματα πολέμου για τους χριστιανούς, ε, Τουρκμένους, Κούρδους, Σιήτες Εάν θέλουμε να είμαστε ακριβείς και συνεπείς με το νομικό πλαίσιο, γιατί πολλοί αναφερθήκατε στο ότι δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά έχει και νομικές επιπτώσεις, αυτό είναι το νομικό πλαίσιο, το ξέρετε. Και μην ξεχνάτε ότι ο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια έδρα στον ΟΗΕ και εργαζόμαστε σε εκείνο το πλαίσιο. Σε εκείνο το πλαίσιο. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις μέσα στο σωστό πλαίσιο που είναι πιο του ΟΗΕ. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι παράλληλα θα πρέπει να δράσουμε πολύ συγκεκριμένα. Όχι μόνο επί της αρχής, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί η περιοχή έχει τα μάτια στραμμένα σε εμά. Και οι μειονότητες κοιτάνε αυτούς που μπορούν να τις υπεραψιστούν. Με λόγια, που και αυτά είναι σημαντικά, αλλά και με πράξεις. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με κάτι που αναφέρθηκε ε, πολύ συγκεκριμένο από κάποιον Ευρωβουλευτή, το θέμα της δικαιοσύνης και της λογοδοσίας. Γιατί όπως είπα και πριν, αλλά θέλω να το επαναλάβω τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την ανεξάρτητη ε, επιτροπή, εξεταστική επιτροπή για τη Συρία που συλλέγει στοιχεία για τις παραβιάσεις που διαπράττονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη των μελλοντικών νομικών ε, δράσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τονίστηκε από εσά, ζήτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παραπέμψει το θέμα της Συρίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα ήθελα λοιπόν να, να πω αυτά ξεκάθαρα. Επίσης να τονίσω και για να κλείσω, γιατί καταλαβαίνω και εγώ ότι έχουμε καθυστερήσει και δεν θέλω να χθοντριβήσω εδώ πέρα, ότι υπάρχουν τρία-τέσσερα πράγματα τα οποία είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας για να προστατεύσουμε τις θρησκευτικέ μειονότητες στη Μέση Ανατολή. Πρώτον, να απελευθερώσουμε τις περιοχές που κατέχει το ΝΤΑΕΣ στο Ιράκ και στη Συρία κυρίως και να τις καταστήσουμε ασφαλείς, να επιστρέψει η κανονική ζωή εκεί. Και εκεί υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια από εμά, στο Ιράκ, γιατί έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση και μπορούν να έχουν μεγαλύτερη δράση, αλλά ελπίζουμε όλο και περισσότερο να συμβεί αυτό και στη Συρία. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για κοινωνίες οι οποίες δεν θα αποκλείουν κανένα. Να ξανά δημιουργήσουμε, θα έλεγα, τις ε, συνθήκες. Γιατί μιλάμε, όπως είπατε και πολλοί από εσά, για κοινωνίες οι οποίες επί αιώνες, αν όχι χιλιάδες χρόνια, ε, ζούσαν μαζί, ειρηνικά και με αμοιβαία κατανόηση. Συζούσαν, συνυπήρχαν και αυτές οι διαφορές ε, πλούτησαν αυτές τις κοινωνίες. Και εδώ μπαίνει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Όχι μόνο πολιτικά, αλλά και ανθρώπινα σημαντικό. Και με εντυπωσίασε που δεν το αναφέρατε σήμερα στη συζήτηση. Γιατί από ό,τι άκουσα από τους χριστιανούς στο Αρμπίλ πέρυσι, το θέμα που συζητάνε περισσότερο είναι αυτό. Ποιο είναι είναι ασφαλέστερο για μας, είναι καλύτερο για μας να μείνουμε στη Μέση Ανατολή ή να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή. Με όλες τις συζητήσεις που γίνονται για την διατήρηση αναδημιουργία του πλουραλισμού σε αυτές τις κοινωνίες της Μέσης Ανατολής. Αυτή είναι μια συζήτηση που κυρίως οι χριστιανοί στις περιοχές αυτές που κατέχει το Ντάεσ στο Ιράκ, αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ έντονες στους χριστιανούς και πιστεύω ότι θα πρέπει να τις ακολουθήσουμε, να τις παρακολουθήσουμε και να τις εντάξουμε στις δικές μας συζητήσεις. Αλλά έχουμε και το καθήκον να τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να επιλέξουν, να δημιουργήσουν ασφαλείς συνθήκες για να ζήσουν στην περιοχή. Γι' αυτό συνδέεται και με αυτό που είπατε κάποιοι ε, από εσά, υποστήριξη των προσφύγων, όλων των προσφύγων και εκείνων που προέρχονται από μειονότητε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματά του, όπου και αν βρίσκονται. Σε οποιοδήποτε μέρο και αν ζουν στην περιοχή. Επίση, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκε και οι προποθέσει να παραμείνουν να επιστρέψουν στι κοινότητέ του, αν το επιθυμούν αυτό, για να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν τον πλουραλισμό των κοινωνιών του. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό καθεαυτό αποτελεί μια αξία, διότι είναι ένα από τα μέρη στον κόσμο όπου διαφορετικά υπόβαθρα, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικές κοινότητες, διαφορές εθνότητες ζούσαν και έδειχναν στον κόσμο ότι να υπήρχε δυνατότητα να συνυπάρξουν. Και πρέπει να κάνουμε το σημαντικό, να σταματήσουμε τις συγκρούσεις, διότι στο κάτω-κάτω αυτό επιτρέπει στις μειονότητες να επιστρέψουν. Και κάτι συμπληρωματικό, κάτι που ακολουθεί. Και κάτι συμβαίνει σε μέρη τα οποία πλησιάζουν σε κάποια κρίση η οποία αυξάνεται. Δηλαδή πρέπει να επενδύσουμε στο να γίνουν ανοιχτές οι κοινωνίες, να υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί, να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, στον πλουραλισμό και στην ένταξη σε αυτές τις χώρες. Παντού, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή να γίνεται αυτό. Εδώ μιλάμε για μια συγκεκριμένη περίπτωση, την περίπτωση του Ντάες ή του ISIS, αλλά όπως είπατε συμβαίνει παντού στον κόσμο αυτό, στην Αφρική, στην Ασία. Μη λησμονείτε τη Λιβύη όπου είχαμε θύματα χριστιανούς διαφορετικών διαφορετικών που σκοτωθήκαν στην Αιθιοπία και στην Αίγυπτο και πρόσφατα και θα πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα. Θα πρέπει να δράσουμε αμέσως, να δώσουμε όλη την υποστήριξή μας ανθρωπιστική καταρχάς να εργαστούμε όσον αφορά τις συνθήκες που επικρατούν για το σεβασμό των μειονοτήτων, την, τον πλουραλισμό και την ένταξη και άμεσα και μακροπρόθεσμα και να καταβάλουμε κάθε διπλωματική προσπάθεια για να τεθεί τέρμα στην κρίση και να νικήσουμε τη μεγάλη πηγή σε αυτή την περίπτωση των προβλημάτων για τις ειδικές μειονότητες στη Μέση Ανατολή που είναι το ΝΤΑΕΣ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση.